Καθίστε παρακαλώ. Γιατί είχαμε ήδη αναβάλει κατά ένα τέταρτο την έναρξη τη απογευματινή μα συνεδρίασης, αλλά ήρθε στο μεταξύ ο υπουργό Εξωτερικών και επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο στην ημερήσια διάταξη, α μην χρονοτριβούμε άλλο. Καταρχήν να σας καλωσορίσω κύριε Υπουργέ. Ξέρουμε ότι η Επιτροπή μας ετοιμάζεται να υιοθετήσει ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα για την κατάσταση στη χώρα σας που, καταχωρεί, που τα καταγράφει τα επιτευχθέντα στοιχεία πρόοδου που μας ικανοποιούν, αλλά έχουμε ακόμα, έχετε ακόμα αρκετά πράγματα να ολοκληρώσετε πριν προσεγγίσετε την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Τα τελευταία χρόνια η χώρα σας κύριε Υπουργέ έδειξε σημαντική κίνηση προς την δημοκρατία και την ελευθερία. Να υπενθυμίσουμε κάποια σημαντικά στοιχεία. Την διακήρυξη της ανεξαρτησίας του 2008, την υιοθέτηση ενός συγχρόνου συντάγματος το Νοέμβριο του 2009 είχαμε τις πρώτες τοπικές εκλογές και την διοργάνωση συνεπώς μιας αποκεντρωμένης δομής δημοκρατικής διακυβέρνησης. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν πρέπει να γνωρίσουμε ωστόσο που ακόμα μπορούν να βελτιωθούν, να συμπενθυμίσουμε ορισμένα τις ε, δυσκολίες τις σχέσεις με την ε, σερβική ε, ε, μειονότητα, την κρίσιμη κατάσταση στο βόρειο κοσφοπέδιο, κάτι που αφορά πιο κοντά εμάς, παραμένει αβέβαιη ακόμα η δραστηριότητα της Eurolex στο Κωσυφοπέδιο, της αποστολής μας. Η διαδικασία μεταρρύθμισης του Κωσυφοπέδιου βεβαίως συνεχίζεται και ο στόχος της δημιουργία ενό λειτουργικού κράτους δικαίου που συμμεριζόμαστε όλοι, είναι κάτι που όλοι ε, θέλουμε και καταγράφουμε τις, τα θετικά βήματα προ την κατεύθυνση αυτή. Χρειάζονται ισχυρά θεσμικά όργανα, τελείω δημοκρατικά. Αυτοί είναι κάποιοι τομείς όπου δεν υπάρχει πλήρης αποσαφήνιση της κατάστασης. Ο δικαστικός τομέας χρειάζονται και άλλες προσπάθειες πέραν αυτών που πρέπει να καταγράψουμε για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Υπενθυμίζουμε την αποστολή Eurolex της Ένωσης που βρίσκεται στο Κωσοπέδιο ακριβώ για αυτό τον σκοπό να ενισχύσει το κράτος δικαίου, να καταπολεμήσει την διαφθορά και να υπάρξει μια αποτελεσματική διαχείριση του δικαστικού συστήματος. Όπως ξέρετε κύριε Υπουργέ, το κοσυφοπέδιο δεν συμπεριλήφθηκε στο πακέτο για την απελευθέρωση των θεωρήσεων που ενδιαφέρει που, που, που, αφορούσε άλλες χώρες της περιοχής. Εμείς ζητήσαμε από την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες για να προχωρήσει γρήγορα προς την φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων και για τους πολίτες της χώρας σας. Un impegno ancora più intenso da... ε, βεβαίως για το σκοπό αυτό χρειάζεται μια εντονότερη δέσμευση από πλευράς της δικής σας χώρας για να πετύχει, για να μπορέσει ο στόχος αυτός να υλοποιηθεί γρήγορα. Με την ευχή αυτή και με πολλές άλλες που μπορούμε να φανταστούμε για το ενδιαφέρον που θα ρίξει η εισήγησή σας. Δεν θέλω να πάρω χρόνο από την συζήτηση. Σας δίνω λοιπόν το λόγο για περίπου 10 λεπτά. Για σας κυρίως, όχι για τους συναδέλφους. Αν θέλετε παραπάνω το πάνω να δούμε. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αλμπερτίνη, χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ξαναβλέπω. By the same token, it's great. Αλλά χαίρομαι που ξαναβλέπω τους πολυάριθμους φίλους εδώ του Κωσυφοπεδίου. Genuinely appreciate the... Γενικώς Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν μου δίνετε ευκαιρία να έχω ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το κοσυφοπαίδιο, σε ποια κατάσταση βρίσκεται και ποιος είναι ο δρόμος μας για το μέλλον. Για τις ε, πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το νεαρότερο κράτος του κόσμου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους ε, βασικούς στόχους και προκλήσεις αυτού του νεοπαγέστερου κράτου στον κόσμο. Και μάλιστα η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η ευρωπαϊκή προοπτική του Κωσυφοπεδίου είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μου. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσά ε, έχουν ε, βαθιά γνώση του τι συμβαίνει στο κοσυφοπαίδιο. Και μια και γνωρίζετε πώς είναι σήμερα το κοσυφοπαίδιο, θα είμαι πολύ σύντομο στις ε, εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, ώστε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων περισσότερο. Γιατί αυτός είναι και ο σκοπός αυτής της συνάντησης, η ανταλλαγή απόψεων. Το κοσυφοπαίδιο συντέλεσε τεράστια πρόοδο κατά τη διετία της ύπαρξής του ως ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους. Προοδεύουμε σταθερά στην οικοδόμηση θεσμών, στην εδραίωση της δημοκρατίας του Κωσυφοπεδίου, που θα θεμελιώνεται σε ένα σύγχρονο σύνταγμα που και πάλι θα στηρίζεται στις ε, υψηλότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Το κοσυφοπαίδιο 24 ώρες το 24ωρο ασχολείται με την εσωτερική εδραίωση της κρατικότητάς του και της διεθνούς ε, εδραίωση της κρατικότητάς του. Εσωτερικά, το κοσυφοπεδίο και οι θεσμοί του κοσυφοπεδίου, το κοινοβούλιο πρώτα απ' όλα της Δημοκρατίας, του κοσυφοπεδίου, κατάφερε μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να υιοθετήσει πολλά νομοσχέδια που ερίζονται στο νέο μας σύνταγμα και στις διατάξεις που προέκυψαν από την ε, συνεκτική πρόταση του πρώην Φιλανδού Προέδρου Μάρτι Ατισάρη. Διεθνώς το Κωσυφοπαίδιο έχει αναγνωριστεί από πολλά έθνη στον κόσμο και ήδη έχει ξεκινήσει διπλωματικές σχέσεις με 30 περίπου χώρες ανά τον κόσμο και ίδρυσε πολλές πρεσβείες και προξενία προκειμένου να εξυπηρετήσει και διμερεί συμφέροντα του κοσυφοπεδίου με τη χώρα υποδοχής της πρεσβείας και του προξενείου, αλλά κυρίως να εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα των υπηκών του κοσυφοπεδίου που διαμένουν στην Αλοδαπή. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι φυσικά ο ύπατος στόχος του κοσυφοπεδίου. Και το κοσυφοπέδιο θα ισχυριστεί ότι έχει ολοκληρώσει την πορεία του από τη στιγμή που θα γίνει δεκτή η χώρα ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας των Ελεύθερων Εθνών. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι η ύψη όθηση και το κίνητρο οποιασδήποτε προσπάθειας που γίνεται στο κοσυφοπαίδιο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να σας διαβιβάσω την εκτίμηση που τρέφει η χώρα μου για την υποστήριξη που πρόσφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον ε, λαό των Κωσοβάρων στη, και στις, στην προσδοκία του για ευρωπαϊκή ένταξη. Και με, έχουμε, διανύουμε κρίσιμους καιρούς. Ε, επίκειται η απόφαση του, του Διεθνούς ε, Ποινικού Δικαστηρίου. Του Διεθνούς Δικαστηρίου, συγγνώμη. Και μπορούμε με τις εξελίξεις που αναμένονται να ισχυριστούμε ότι ε, έπονται κρίσιμοι καιροί που χρήζουν και κρίσιμων αποφάσεων. Μερικές φορές θα είναι δυσχερείς αυτές οι αποφάσεις, αλλά θα είναι και απαραίτητες αν θέλουμε να προχωρήσουμε με ασφάλεια και ως υγιές κράτος και ατομικά μεμονωμένα ως ε, χώρα των Δυτικών Βαλκανίων αλλά και συλλογικά ως περιφέρεια ζώνη των Δυτικών ε, Βαλκανίων. Το Κωσυφοπαίδιο έχει αναλάβει τη δέσμευση, την πάγια δέσμευση να υλοποιήσει το στόχο της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τον υλοποιήσει μάλιστα εκ παραλίλου με το στόχο της ε, δημιουργίας στενών και αγαστών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες και την υλοποίηση της περιφερειακής συνεργασίας. Έχουμε εξαιρετικές ε, σχέσεις με όλες τις γειτονικές μας χώρες, τις όμορες χώρες και επιδιώκουμε ομαλές σχέσεις και με την ε, Δημοκρατία της Σερβίας. επιμένουμε να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μας με τη Δημοκρατία της Σερβίας γιατί το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και θα πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε όριμοι για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αναζητώντας και εντοπίζοντας πιο επικοδομητικούς τρόπους ε, συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο. Instead of throwing up Αντί λοιπόν να ορθώνουμε διπλωματικά κολλήματα και προσκόμματα στο δρόμο του κωσυφοπεδίου, πιστεύω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ώστε η δημοκρατία της Σερβίας ε, να δεχτεί μια διαφορετική κατεύθυνση, μια διαφορετική πορεία, την πορεία της συνεργασίας, χάρη της περιφερειακής ειρήνης, αλλά και χάρη της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων το να εγείρονται όλο και περισσότερα διπλωματικά προσκόμματα και σκόπελοι στο δρόμο της ε, εδραίωσης, της διεθνούς εδραίωσης της ε, κοσοβάρικης ε, κρατικότητας, είναι σαν να προσπαθεί κανείς να διευρύνει το φάσμα της αντιπαράθεσης μεταξύ της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Δημοκρατίας του Κωσυφοπεδίου. Θα πρέπει να διερευνήσουμε διαφορετική κατεύθυνση, να μειώσουμε το φάσμα της αντιπαράθεσης και να διευρύνουμε τη συνεργασία σε πολλά ζητήματα που μας ενδιαφέρουν και τις δύο πλευρές. Χαιρόμαστε για την επέκταση του οδικού χάρτη για την απελευθέρωση των θεωρήσεων για την Αλβανία και τη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Το συντομότερο δυνατό. Ταυτόχρονα όμως ζητούμε έναν σαφή κατάλογο με συγκριτικούς κανόνες και καθήκοντα που θα πρέπει να επιτελέσει το κοσυφοπαίδιο, ώστε και η χώρα αυτή να λάβει τον οδικό χάρτη το συντομότερο δυνατό. Γιατί είναι κολοσιαίο λάθος να παρεμποδιστεί ή να παρακολουθεί αυτή ε, η διαδικασία για το κοσυφοπαίδιο της απελευθέρωσης των θεωρήσεων και να ε, καθυστερήσει πολύ περισσότερο από ό,τι για τις δύο άλλες χώρες. Φυσικά και το κοσυφοπαίδιο έχει πολλά καθήκοντα να επιτελέσει και μάλιστα ήδη διαπραγματευόμαστε συμφωνίες επανεισδοχής με πολλές ε, κοινοτικέ χώρες. Ήδη έχουμε υπογράψει τρει τέτοιες συμφωνίες με τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Αλβανία. Και μάλιστα ολοκληρώσαμε διαπραγματεύσεις με Αυστρία και Νορβηγία και απομένει ένας γύρος διαπραγματεύσεων με την Αυστρία. Είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε οποιουσδήποτε συγκριτικούς κανόνες επιβάλλεται. Να είστε απαιτητικοί απέναντι στο κωσυφοπέδιο, να είστε αυστηροί μαζί μας. Δώστε μας όμως έναν σαφή κατάλογο και μία σαφή ιδέα για το χρονοδιάγραμμα. Ούτε εμείς, αλλά ούτε και εσείς φαντάζομαι θέλετε να μας δείτε σε μια δυσάρεστη κατάσταση. Γιατί το Σύνταγμα του Κωσυφοπεδίου προβλέπει διπλή ηθαγένεια και δεν θέλουμε να σπεύσουν οι πολίτες μας, οι υπηκοοί ε, να, βγάλ, να εκδώσουν σερβικά, βοσνιακά ή αλβανικά διαβατήρια μόνο και μόνο για να υποφεληθούν από την κατάργηση των θεωρήσεων. Πολύ ευγενικά ο κύριος ε, πρόεδρος μου επισημαίνει την πίεση του χρόνου. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την ε, προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Σίγουρα στη συνέχεια της συζήτησης θα μπορέσετε να επεκταθείτε στα θέματα που αφήσετε εκρεμή. Ξεκινούμε με την κυρία Λούνα Τσεκ που έχει τρία λεπτά ως εισηγήτρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ τον Υπουργό που ήρθε και μας έκανε αυτό, αυτή την εντυπωσιακή εισήγηση. Χαίρομαι που σα συναντώ σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και όχι μόνο στο γραφείο μου ή τέλο πάντων σε άλλου χώρου του Κοινοβουλίου. Ξέρετε ότι προετοιμάζουμε την έκθεση. Είχαμε μια πρώτη συζήτηση στο Κοινοβούλιο ήδη. Εκτιμώ αυτό που είπατε και αυτό που ακούω εδώ στις τρεις, εβδομα... στις τρεις επισκέψεις που έχω μέχρι τώρα κάνει στο Κοσφοπίδιο τελευταία, την περασμένη εβδομάδα. Μας είπατε να είσαστε απαιτητικοί μαζί μας. Το εκτιμώ αυτό, ε, διότι όπως αναφέρθηκε υπάρχουν όντω πολλά πράγματα που πρέπει να κάνετε εσείς και η κυβέρνησή σα, Θέλω ωστόσο από πλευρά μου να επιβεβαιώσω και εξ πολλών στο Κοινοβούλιο, πολλού ε, βουλευτές, την υποστήριξή μας προς την πορεία σας προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Είπατε και εσείς, είναι σημαντικό να μην είναι οι πολίτες της χώρας σας απ' έξω ενώ όλοι γύρω σας μπορούν να ταξιδέψουν και να μην οδηγηθούν οι πολίτες του να πάρουν υφαγένειες άλλων χωρών εγώ σας υποστηρίζω, εμείς σας υποστηρίζουμε και αυτή η προσέγγιση είναι νομίζω μια προσέγγιση που ακολουθούμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε, είμαι μεταξύ αυτών που παλεύουν και αγωνίζονται να αναγνωρίσουν και τα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης στην χώρα σας το συντομότερο δυνατό. Ξέρω ότι έχουμε χρόνο μπροστά μας. Ας μιλήσω. Θα ήθελα να μιλήσω για κάποια από τα σημαντικά θέματα που πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να τα θέσουμε σαφώς στι σχέσει μεταξύ Κοινοβουλίου, Ένωση και τη χώρα σα. Είπατε κι εσεί ο ίδιο ότι το κράτο δικαίου, η εγκαθίδρυση πλήρω λειτουργών, λειτουργών των θεσμών είναι ουσιαστική και για εσά. Συμφωνώ μαζί σα. Κάτι που θέλω να ρωτήσω. Πρόσφατα έγινε ένα σχηματισμό στην κυβέρνηση. Υπάρχουν νέοι υπουργοί στον τομέα της παιδείας και της υγείας. Το μίσο που χρειάζεται μεγάλη δουλειά στη χώρα σας για να έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα ανοιχτό σε όλους και σε ένα σύστημα υγείας καλό για όλους. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται στον τομέα αυτό. Κάτι άλλο που με εξέπληξε θετικά όταν είχα πάει την περασμένη εβδομάδα στην Πρίστινα. Η, τα, η σήμανση στους δρόμους είναι σε τρεις γλώσσες. Αλβανικά, σερβικά και τουρκικά. Γλώσσες που μιλούν. Υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια στην ε, χώρα σας να ενισχυθεί η πολυγλωσία, να μαθαίνουν σερβικά οι Αλβανοί, αλβανικά ή Σέρβοι κλπ. Um, there is one thing that you know has been very much over the last weeks. Κάτι που... Κύριε Πρόεδρε, μου δίνετε ένα λεπτό ακόμα. Κάτι που επικρίθηκε την περασμένη εβδομάδα ήταν η διακοπή των αναμεταδοτών ε, εταιριών σερβικών ε, κινητής τηλεφωνίας. Κάτι που ήταν σοκ για όλους όσοι ε, είχα πάει στο Στρίψ την περασμένη εβδομάδα και είχα μιλήσει με δημάρχους. Αυτό πραγματικά που κάνετε έπληξε αυτούς που ήθελαν να ενισχύσουν τις σχέσεις ε, των δύο κοινοτήτων. Ξέρω ότι κάποιε από τι κάποιες από εταιρείε δεν είχαν άδεια και ότι θέλετε ε, να, να, να, το αλλάξετε αυτό. Αλλά θα έπρεπε να μπορούν όλοι οι πολίτες του Κόσοβο να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν σωστά τηλεφωνήματα. Μεταφορές τώρα. Η κυβέρνησή σα αποφάσισε να δώσει 700 εκατομμύρια ευρώ στον αυτοκινητόδρομο προς την ε, Αλβανία που είναι 20% του ΑΕΠ της χώρας σας. Πιστεύετε ότι αυτό το ποσό είναι το, το, το, τα κονδύλια αυτά είναι ο καλύτερος τρόπος χρησιμοποίησης τους ή υπάρχουν και άλλοι καλύτεροι. Ευχαριστούμε κύριε Λούνατσεκ. Ήθελα να σας να περιορίσω την χυμαρόδη ε, ικανότητά σας να, να μιλήσετε για να αφήσω και σε άλλους συναδέλφους το δικαίωμα να παρέμβουν. Ε, ο κύριος Κούκιν, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον προσκεκλημένο. Να σας ευχαριστώ που ε, ήρθατε εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Δύο θέματα θα με ενδιαφέραν. Αναφέρατε ήδη το πρώτο από αυτά, σύντομα, τη σχέση σας με τη Σερβία. Η ερώτησή μου αφορά την περιφερειακή συνεργασία στα Βαλκάνια, διότι όλοι γνωρίζουμε την σημασία αυτού του είδους συνεργασίας είναι η καλύτερη προετοιμασία για το μέλλον της χώρας σας ως προς ε, την ε, προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη παρατήρηση, όσον αφορά τα πέντε κράτη-μέλη, που μέχρι στιγμής δεν έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του κοσφοπεδίου. Ακούμε μερικές φορές εκκλήσεις εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τις χώρες αυτές να αναγνωρίσουν το κοσυφοπέδιο. Αυτό δεν έχει αλλάξει τη θέση τους. Όταν Μιλήσατε για την ε, εξάλληψη των ε, διεθνών μπλοκ. Ε, Ελπίζω να μην αναφερόσασταν στι πέντε αυτέ χώρε, γιατί η χώρα μου, η Σλοβακία, έχει δείξει ότι και χωρί επίσημη αναγνώριση μπορούμε να έχουμε χρήσιμο διάλογο. Μύροσλαβ Λάιτσεκ από τη Σλοβακία έχει αποδείξει ότι είναι δυνατός ο διάλογος με τη χώρα σας. Ωστόσο, θα ήθελα να ακούσω τις ειλικρινές σας τις ειλικρινείς σας παρατηρήσεις για το θέμα αυτό, το θέμα δηλαδή των σχέσεων του κοσφοπεδίου με τις πέντε αυτές χώρες. Ο κύριος και ο ηγητής για τους σοσιαλιστές. Τρία λεπτά και λιγότερα ίσως, λέει ο μιλητής. Καταρχάς, καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι είπατε σήμερα λόγια που όλοι μπορούμε να συμμεριστούμε. Ανήκω σε εκείνους που θεωρούν ότι είναι αναγκαία η ένταξη της χώρας σας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και γι' αυτό θέλω να πω κάποιες παρατηρήσεις με τη μέγιστη δυνατή ειλικρίνεια. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι έγιναν βήματα μπρος στην θεσμική και δημοκρατική σταθεροποίηση. Το είδαμε αυτό με τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, τις οποίες είχα την ευκαιρία να ήμουν παρόν και να τις παρακολουθήσω εκ του σύναγκης. Επιπλέον, η παγίωση και στερέωση των θεσμικών αυτών πυλών ήταν προϋπόθεση για την προσέγγιση της χώρας σας στην, προς την Ευρώπη και εμείς είμαστε εδώ για να ενθαρρύνουμε τη διαδικασία αυτή. Ωστόσο υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμα. Έχετε δίκιο όταν λέτε δώστε μας ένα χρονοδιάγραμμα. Ε, πιστεύω ότι έχετε δίκιο όταν μιλάμε για θεωρήσεις, για παράδειγμα. Πιστεύω ότι σωστά λέτε πρέπει να εντοπίσουμε έναν δρόμο για μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση. Υπάρχει ωστόσο ένας κατάλογος που σας δόθηκε κατά κάποιο τρόπο και σταματώ σε δύο θέματα που θεωρώ ουσιαστικά για να στερεώσουμε την, τον εκδημοκρατισμό και την προσέγγιση της στην Ευρώπη. Πρώτον, λειτουργία των θεσμών, ιδίω της δικαιοσύνης. Υπάρχει ανάγκη πιο βαθιών μεταρρυθμίσεων για να αποκτήσει η δικαιοσύνη πολύ πιο στέρεα βάση. Δεύτερο ζήτημα. Ένα πρόβλημα που προφανώς ε, δεν αφορά μόνο τη χώρα σας και άλλες αφορά αλλά που είναι ιδιαίτερα εμφανές εκεί και σχετίζεται με θέματα διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος που ουδόλως έχουν επιληθεί. Και αυτά είναι θέματα που σχετίζονται με την αποστολή της Eurolex στο Κοσφοπέδιο. που ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει στην δημοκρατική σταθεροποίηση. Μήπως θεωρείτε χρήσιμο και αναγκαίο στους δύο αυτούς τομείς να γίνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια, μια πιο σοβαρή προσπάθεια από τη χώρα σας ακριβώς, ούτως ώστε ο κατάλογος που ζητάτε και το πρόγραμμα που αναφέρετε να μπορέσουν να συμφωνηθούν το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παντσέρη. κύριος Κάτσιν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Eh, Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι ιδιαίτερος για την παρουσία σας στην Επιτροπή μας και είμαι ιδιαίτερη υπερήφανος για τη συμβολή της Γιούλεξ στην ε, ανοικοδόμηση των θεσμών στο Κωσυφοπαίδιο. Χθες συναντηθήκαμε με Αλβανούς βουλευτές και πιστέψτε με ότι το Κεντρικό θέμα της συζήτησής μας ήταν η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η πάταξη της διαφθοράς και μάλιστα ιδιαίτερα σε υψηλά κλιμάκια και σε στελέχη της κυβέρνησης. Υπάρχει, υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα στις σχέσεις της χώρας σας με τη Γιούλεξ. Τι προσπάθειες θα πρέπει να γίνουν για να παταχθεί η διαφθορά. Η κυρία Τσέκ. αναφέρθηκε στα προβλήματα που έχουν οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Άλλο όμως να απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλο να καταστρέφονται κινητά. Δεν είναι καλύτερο να κλείνουν αυτές, να απενεργοποιούνται αυτές οι συσκευές αντί να καταστρέφονται, γιατί έτσι ε, δημιουργείται περιθώριο διαλόγου με το Βελεγράδι δημιουργείται δυνατότητα ανέβρεση λύση που θα εξυπηρετεί και τι δύο πλευρέ, και τη σερβική μειονότητα και τη Σερβία. Αλλά και τον αλβανικό πληθυσμό του Κωσυφοπεδίου. Και τελευταία μου ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Στις 2 Ιουνίου θα λάβει η χώρα στο Σαράγεβο η συνδιάσκεψη για τα Βαλκάνια. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει για το κατά πόσο θα παραστούν εκπρόσωποι όλων των χωρών. Ερωτώ, εσείς θα δώσετε το παρόν στο Σαράγεβο, κύριε Υπουργέ. Ο Λέζινγκ, δύο λεπτά. Η κυρία Λέζινγκ, δύο λεπτά. Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω και να σας παρακαλέσω να απαντήσετε στην εξή ερώτηση. Από την αλβανική πλευρά στο Κόσοβο ε, Γίνονται όλο και πιο πολλές ε, διαμαρτυρίες για την ε, παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ο Ήλεξ Κόσοβο έχει προσφύγει κατά των διαμαρτυρουμένων των διαδηλωτών με τα κρυγόνα. Εσείς πώς το βρίσκετε αυτό, βρίσκετε αναλογικά τα μέτρα και κύριε Υπουργέ, δεδομένων των αυξανόμενων διαμαρτυριών η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΚΑΦΟΡ έχει ξεκινήσει ασκήσεις με την ε, k για να βελτιώσει την δυνατότητα ε, ε, καταστολής των διαδηλώσεων. Πρόσφατα είχαμε ήδη τρεις τέτοιες καταστολές. Εσύ πώς κρίνετε την εξέλιξη αυτή. Το 79% του του πληθυσμού του Κωσόβου λόγω της, καλής, ε, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης είναι τεθμένα να συμμετέχουν στις ε, διαδηλώσεις. Το Κωσυφοπαίδιο έχει ένα από τα πιο φιλελεύθερα καθεστώτα εμπορίου στον κόσμο, λέει η Παγκόσμια Τράπεζα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα μέτρα οδηγούν σε βελτίωση ή σε επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης. Ο Χέλμουτ Κούν, σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής, είχε ζητήσει να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη ε, και μιλούσε για προτεκτοράτο όσον αφορά την ε, λύση Αχτισάρη. Έλεγε ότι δεν είναι πραγματικό καθεστώς ανεξαρτησίας. Είναι Ε, αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ε, καταργήσει οποιοδήποτε, οποιοδήποτε κομμάτι νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απολύσει οποιονδήποτε υπουργό. Ποιο αποφασίζει το Κόσοβο. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τάλερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Κόσοβο ως κράτος βασίζεται στην προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου από την πλειοψηφία του πληθυσμού, κάτι το οποίο το καθεστώς του Μιλόσεβιτς δεν ήθελε να πετύχει να κάνει. Πιστεύω ότι η στάση σας αυτή σας υποχρεώνει ηθικά να δείξετε τι μπορείτε να κάνετε τώρα που γίνετε ανεξάρτητοι, να δείξετε πώ μπορείτε να αναπτύξετε τη δημοκρατία στο πεδίο, να προωθήσετε τα δικαιώματα των, του ανθρώπου, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, να χτυπήσετε τη διαφθορά και να, ε, να εκμεταλλευτείτε καλύτερα το, τις δυνατότητες της νεολαίας σας. Αυτά είναι τα κριτήρια πάνω στα οποία θα κρίνουμε το κουσιφοπέδιο. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι σας αναγνώρισαν, εγώ τουλάχιστον. Η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη και σχετίζεται με αυτό που ρώτησε ο συνάδελφος κ. Κουτσίν για την σύνοδο του Σαράγεβο που οργανώνεται υπό την αιγίδα της Ισπανικής Προεδρίας. Καλή επιτυχία στην σύνοδο αυτό. Νωρίτερα χρειάστηκε να αγνοήσω την αδιαφορία που έδειξε η Ισπανική Προεδρία πριν από 1,5 μήνα όταν μια αντίστοιχη διάσκεψη για τα Δυτικά Βαλκάνια οργανώθηκε στο, στη Σλοβενία, στο, στο ε, Στην συνάντηση εκείνη ήταν παρόντες όλοι οι επικεφαλείς των κρατών μελών των Δυτικών Βαλκανίων με μία εξαίρεση μιας χώρας. Ποια είναι η θέση σας σήμερα, ποια είναι η θέση της κυβέρνησής σας για την διάσκεψη του Σαράγεβο υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμού που θα επιτρέψει να συμμετάσχουν και οι δύο χώρες ταυτόχρονα, η Σερβία και το Κωσυφοπέδιο. Ευχαριστώ. Τον πρώτο γύρο τον ολοκληρώνει ο κύριος Σαλαφράνκα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Το πρωί ο εκπρόσωπος της ΥΠΑ της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική μας ενημέρωσε διεξοδικά για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και μάλιστα ανέπτυξε με λεπτομέρεια τα τέσσερα σημεία της αποστολής Γιούλεξ στο Κωσυφοπαίδιο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Ο κύριος Χισένη γνωρίζει από που κατάγομαι, γνωρίζει τη θέση της Ισπανίας για το Κωσυφοπαίδιο και η μοναδική ερώτηση που έχω να το απευθύνω είναι ποιες είναι οι σχέσεις του Κωσυφοπεδίου με την ε, ασκούσα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισπανία. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Αν μπορέσετε να τηρήσετε το δεκάλεπτο, θα σας ήμουν ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ λογικά τα ερωτήματα όλα αυτά και οι παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ όλους. Όσον αφορά την ε, ε, την αλλαγή της κυβέρνησης είχε στόχο να βελτιώσει τη διακυβέρνηση σε κάποιες από τις ε, κρίσιμες περιοχές. Η αναδιάφρωση αυτή έγινε πριν λίγο καιρό για να... και θέλουμε να δώσουμε στους νέους υπουργούς λίγο περισσότερο χρόνο ε, για να κρίνουμε εάν ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους και αν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες. σχετικά με την συμμετοχή του στην κυβέρνηση. Όσον αφορά τις γλώσσες, η πλειοψηφία της αλβανικής, ε, του αλβανικού πληθυσμού του, Κωσόβου, του ε, ξέρει να μιλάει σέρβικα και αυτό είναι πολύ καλό. Ε, φοβάμαι ότι δεν μπορώ να πω το ίδιο για τους Σέρβους του Κωσοφοπεδίου. Αλλά βλέπουμε να υπάρχει πρόοδος και σε αυτό το μέτωπο και σίγουρα Η εκμάθηση της γλώσσας των άλλων εμπλουτίζει τους ανθρώπους. Εμείς ως κυβέρνηση ενθαρρύνουμε το να γίνεται αυτό. Φυσικά, κάποια θέματα χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες στο κοσυφοπαίδιο με πρόσφατες αναμνήσεις των γεγονότων ε, του πρόσφατου πολέμου στο Κοσφοπέδιο. Ξέρω ότι για κάποιους πολίτες του, ε, του Κοσφοπεδίου η απομάκρυνση των κεραιών παράνομων ε, παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ήταν σοκ και δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Σας διαβεβαιώ ότι δεν έγινε η παραμικρή πολιτική κίνηση, δεν υπήρξε το παραμικρό πολιτικό κίνητρο πίσω από τη δράση αυτή. Η μόνη πρόθεση ήταν η αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Η απομάκρυνση παρανόμων παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Οι ίδιες επιχειρήσεις που ενεργούσαν παράνομα στο κοσυφοπαίδιο είναι ευπρόσδεκτες να διαπραγματευτούν εμπορικές, νόμιμες εμπορικές συμφωνίες και συμφωνίες περιαγωγής με τους νόμιμους παρόχους υπηρεσιών στο, κοσο, στο κοσοπέδιο όπως είναι η ΥΠΚΟ και άλλοι. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε για να, ε, για να περιορίσει τις, ε, τα προβλήματα που είχαν οι πολίτες του Κοσμοπεδίου ως αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής. Ε, συνεχίζεται η διανομή δωρεάν καρτών SIM προς όλους τους πολίτες του Κοσφοπεδίου που επηρεάστηκαν ε, από την ενέργεια αυτή της ε, ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής για τις τηλεπικοινωνίες. Όσον αφορά τον αυτοκινητόδρομο προς την Αλβανία, ομολογώ ότι είναι πολύ ακριβό έργο, αλλά τελικά απαραίτητο για το κοσφοπέδιο. Για την καλύτερη πρόσβαση από το κοσφοπέδιο προς τη θάλασσα. Μακροπρόθεσμα είναι ένα απαραίτητο έργο, εμπορικά βιώσιμο και ε, ιδιαίτερα σκόπιμο. Φυσικά θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό μας, αλλά θα πρέπει να κατασκευάσουμε τέτοια έργα όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι, ε, τα νέα ε, ε, εργοστάσια θερμότητας και ενέργειας για να θέσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ε, για μακροπρόθεσμη ε, αποκατάσταση και ανάπτυξη της οικονομίας. Κύριε Κούκαν, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ε, όσον αφορά τις σχέσεις με τη Σερβία και τη συμμετοχή του κοσμοπεδίου σε περιφερειακές πρωτοβουλίες. Είναι ζωτική σημασία στα θέματα αυτά. Το κοσμοπέδιο θέλει να συμμετάσχει και επιμένει σε αυτό. Επειδή άκουσα και άλλες ερωτήσεις σχετικά με αυτό, θα, κλείσω, θα συνεχίσω την απάντηση για το θέμα αυτό αργότερα. Όσον αφορά την ε, αναγνώριση από τα πέντε τελευταία κράτη-μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους φίλους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα το κοσμοπέδιο για να το κάνουν αυτό. Διότι είμαστε πεπισμένοι ότι αναγνωρίζοντας το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος, βοηθάτε εξίσου και τη Σερβία και το κοσφοπέδιο. να μην προσποιούμαστε ότι η μία αναγνώριση βοηθάει τη Σερβία. Είμαι βέβαιο ότι τα πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσμοπέδιο δεν λένε αυτό. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με τα κράτη που δεν μας έχουν αναγνωρίσει για να τους παράσχουμε οτιδήποτε μπορεί να τους βοηθήσει να εξετάσουν τη δυνατότητα ε, αναγνώρισης και να λάβουν σχετική απόφαση. Το κάνουμε αυτό σε διάφορα επίπεδα. Και να φτάσω στην ερώτηση του κυρίου Σαλαφράνκα. Τι κάνει το κοσμοπέδιο και πώς. Και τι επαφές έχουμε με την Ισπανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούμε να βρούμε διάφορους τρόπους επικοινωνίας μερικές φορές σε διεθνείς διασκέψεις και σε άλλα μέρη, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι δεν υπάρχει ένα ε, κανάλι τακτικής επικοινωνίας. Όσον αφορά το δικαστικό σύστημα, Αυτός είναι ένας τομέας στο κοσυφοπαίδιο, κύριε Παντσέρη, στον οποίο δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Η μεταρρύθμιση του τομέα αυτού είναι ζωτική σημασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και ε, είμαστε αποφασισμένοι να δούμε αποτελέσματα στον τομέα αυτό. Είμαστε αποφασισμένοι όχι μόνο να ε, παράσχουμε ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο φυσικά είναι απαραίτητο και αποτελεί προπόθεση για την επιτυχία μας ε, στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθορά. Είμαστε, δεσμευόμαστε ε, να έχουμε αυτά αποτελέσματα στον τομέα αυτών. Και είμαι βέβαιος ότι θα το δείτε αυτό πολύ σύντομα. Πρόκειται για νέο κράτος. Δύο χρόνια ζωής έχει. Έχουμε πολλά στο πιάτο μας. Και φυσικά δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε τόσα θέματα, τόσες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ένα νέο κράτος. Αλλά κανείς δεν θα πρέπει να αμφισβητήσει την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα. Υπάρχουν πολλοί αρνητικά φαινόμενα ε, στην κοινωνία μας και αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε πρώτα, θα τους δώσουμε προτεραιότητα. Κύριε Κάτσιν. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά. Όσον αφορά την απομάκρυνση των κεραιών, μπορώ μόνο να τονίσω ότι το μόνο κίνητρο για την πράξη αυτή ήταν η αποκατάσταση του κράτους δικαίου σε όλα τα μέρη της χώρας μας, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για επιτυχία σε πολλά άλλα μέτωπα. 2 Ιουνίου και διάσκεψη του Σαράγεβο διάσκεψη κορυφή. Η διάσκεψη του Γκίμνικ στην Πράγα ήταν εξαιρετικό πλαίσιο που μας έδωσε τη δυνατότητα να συμμετάσχουν όλοι οι Υπουργοί Εξωτερικών από τα Δυτικά Βαλκάνια σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Εφόσον εφαρμοστεί το ίδιο στο Σαράγεβο, το Κωσυφοπαίδιο είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί, να συμμετάσχει. Και θα θέλαμε να δούμε όλο τον κόσμο στο Σαράγεβο. το Gimnik είναι ένα άτυπο πλαίσιο και δεν βλέπω κανένα λόγο να μην συμμετάχει οποιοδήποτε από τους, ε, από τους εμπλεκόμενους στο πλαίσιο αυτό. Είναι αλήθεια, κυρία Λέζινγκ, ότι γίνονται διαδηλώσεις σε διάφορα μέρη κατά καιρού στο Κόσοβο. Το Κοσφοπέδιο ως νέα δημοκρατία είναι αποφασισμένο να αναπτυχθεί σε μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία. Το δικαίωμα διαδηλώσεων είναι δικαίωμα το οποίο προσυπογράφουμε απόλυτα. Ταυτόχρονα, προσυπογράφουμε και στο νόμο και την τάξη. Μονάδες ελέγχου των πληθών, είτε μιλάμε για το Ulex, το k e ή την αστυνομία του Κοσμοπεδίου. Είναι απόλυτα αρμόδιες να διασφαλίσουν το σεβασμό του νόμου και της τάξης. Δεν είμαστε προτεκτοράτο, καλέσαμε το Ιούλεξ να έρθει σε μια ανεξάρτητη χώρα για να υποστηρίξει τα θεσμικά όργανα του Κωσόβου. Στους τομείς ε, της αστυνομίας και του δικαστικού συστήματος. Καλωσορίζουμε την παρουσία αυτή και κάθε μέρα συνεργαζόμαστε πιο στενά για να αντιμετωπίσουμε τις πολλές προκλήσεις στον τομέα της αστυνόμευσης και του δικαστικού συστήματος. Η διεθνής παρουσία στο Κωσυφοπαίδιο βασίζεται στην πρόταση Αχτισάρη. Πρόταση ε, που έχει εγκριθεί απόλυτα από το Κοινοβούλιο του Κοσφοπεδίου. Πρόταση που ε, ταιριάζει απόλυτα με το Σύνταγμά μας. Η παρουσία της Ιούλεξ, της ICO στο Κοσμοπέδιο δεν είναι τίποτα περίεργο διότι βασίζεται στη Συμφωνία Αχτισάρη. Και η παρουσία αυτή βασίζεται σε απόφαση της ε, κυρίαρχης ε, αρχής του κοσφοπεδίου. Κύριε Τάλερ, σας ευχαριστώ για την παρατήρησή σας και για τις ερωτήσεις σας. Επαναλαμβάνω. Πολλοί από εμά. Εργαζόμαστε για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των υποστηριχτών του κοσφοπεδίου εμείς που κατέχουμε αξιώματα. Όχι απλά έτσι για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες, αλλά και για να μετατρέψουμε τη χώρα μας σε μια δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα με ευημερία. Το Κωσυφοπαίδιο αποτελεί μέρος της Ευρώπης και νιώθει πολύ έντονα ότι είναι μέρος της Ευρώπης. Ο χάρτης Ευρώπης δεν, δεν μπορεί να συμπληρωθεί να, να ολοκληρωθεί χωρίς το κοσμοπέδιο. Γι' αυτό είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχει στους ανθρώπους του κοσφοπεδίου ε, μια απτή ευρωπαϊκή προοπτική, πολύ απτή. Ελπίζω να σεβάστηκα το χρόνο, αλλά να επανέλθω στο στο, στη διάσκεψη κορυφή του, του Σαράγεβο. Ναι, σε μια σειρά πρόσφατων συναντήσεων που είχα με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ιταλίας, τον Φραγκοφρατίνη της Γαλλίας, τον Μπέναρ Κούσνερ χθε. και μια εξαιρετική συνάντηση που είχα σήμερα το απόγευμα με τον Επίτροπο Στέφαν Φίλε παρουσίασα τη συνένεση του Κοσμοπεδίου να συμμετάσχει στη διάσκεψη κορυφής του Σαραγεύου. Εφόσον βέβαια οι διοργανωτές ε, μας διαβεβαιώσουν ότι θα εφαρμοστεί το φορμά γκίμνιχ Πράγας διότι το πλαίσιο αυτό παρέχει για όλους τους συμμετέχοντες ασφάλεια. Κάθε, ε, ο καθένας μπορεί να συμμετέχει με αξιοπρέπεια στο πλαίσιο αυτό. Προσβλέπουμε λοιπόν ε, στην συνάντηση του Σαράγεβο ακόμα περισσότερο προσλέπουμε στην ουσία της διάσκεψης του Σαράγεβο. Και το κοσφοπέδιο, πολύ σωστά, περιμένει και στο Σαράγεβο να δοθεί μια σαφής προοπτική για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σας ακούσαμε με πολύ ενδιαφέρον, άρα για να σας πω την αλήθεια. Όχι απλά δεν τηρήσετε, αλλά ξεπεράσετε κατά πολύ το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας. Βέβαια, τα επιχειρήματα, τα θέματα που αναφέρετε, απαντούσαν στα ερήματα. Ο κ. Σεβερίν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Χισένη, σας ξέρω πολλά χρόνια πάντα υποστηρίζεται το, την υπόθεση του λαού σας. Σήμερα, ωστόσο, για κάποιου από εμά είστε υπουργό εξωτερικών ενό αναγνωρισμένου κράτου, ενώ για άλλου είστε ο εκπρόσωπο των κοσοβάρικων προσδοκιών. Όλοι είμαστε έτοιμοι, βέβαια, να βοηθήσουμε τη χώρα σα στον στόχο να πετύχετε τι προσδοκίε αυτέ. Να σας πω ωστόσο ότι η αναγνώριση δεν φτιάχνει το κράτος, το ανάποδο. Ένα πολιτικά οργανωμένο αφ, ε, ε, που, που στηρίζει τον εαυτό του κράτος αποτελεί προϋπόθεση αναγνώρισης. Και από την άποψη αυτή η δουλειά που πρέπει να κάνετε είναι ακριβώς εσωτερική κύριος, μέσα στη χώρα σας. Προφανώς ωστόσο αν δεν υπάρξει μία σύγκληση των απόψεων για την αναγνώριση του κράτους, τίθεται επαμφιβόλο το μέλλον σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας, το μέλλον σας είναι να, γίνει, να γίνετε μέλος της Ένωσης. Και η ερώτησή μου είναι εξή. Για να υποστηρίξουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας σας, χρειαζόμαστε ένα νέο πολιτικό πλαίσιο στην περιοχή των Βαλκανίων. Το θέμα δεν είναι μόνο η συνεργασία, αλλά μια νέα δυναμική, ένα νέο πλαίσιο. Διότι χωρίς να έχετε καλές γειτονικέ σχέσεις με άλλους, δεν μπορεί να έχετε μέλλον στην Ένωση. Έχετε μια εικόνα του τι θέλετε να κάνετε. Προσπαθείτε να αλλάξετε το πλαίσιο στα Δυτικά Βαλκάνια, ώστε να μας επιτρέψετε να ξεπεράσουμε τις εφυλάξεις αυτών που σήμερα σας αναγνωρίζουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάγγελ, δύο λεπτά. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Στην σεβάσμη αυτή συνέλευση. Περιμένετε να σας αναγνωρίσουν όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Είμαι βέβαιος ότι δικαιολογημένα το περιμένετε αυτό για τους λόγους που ανέφερε ο συνάδελφος κ. Σεβερίν. Πρέπει να σας πω ότι καταλαβαίνω καλύτερα τα αισθήματα και τις δραστηριότητες της Σερβίας που θέλει να εμποδίσει την αναγνώριση. Περισσότερο το καταλαβαίνω αυτό παρά τη συμπεριφορά των κρατών εκείνων που δηλώνουν ότι δεν είναι έτοιμα να αναγνωρίσουν τη νέα πραγματικότητα που προέκυψε στην περιοχή και δεν το παραδέχονται. Βεβαίω, λέω ότι καταλαβαίνω καλύτερα τη θέση της Σερβίας. Θέλω ωστόσο να πω ότι καλό θα ήταν να είσαστε ανοιχτοί και στους δημάρχους της ε, σερβικής κοινότητας. Δείξετε ότι ε, θέλετε να ε, βοηθήσετε συμπεριλαμβάνοντας τους Σέρβους στο ψηφοδέλτιο των φιλελεύθερων. Καλή ιδέα και χρήσιμη. Προσέξτε ωστόσο το εξής. Η εγκληματικότητα και η προσπάθεια καταπολέμησης της εγκληματικότητας πρέπει να προσεχτούν περισσότερο. Και μην ξεχάσετε και την αντιμετώπιση των Ρωμά. Ο κύριος Αγκουράκης, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ε, δυστυχώς δεν μπορώ να προσφωνήσω τον ε, κύριο Χισένη με τον τίτλο που τον προσφώνησαν όλοι οι υπόλοιποι που μιλήσανε, γιατί κατά τη γνώμη μου εξακολουθεί να ε, εκπροσωπεί μια οντότητα η οποία είναι απόσχηση από τη Σερβία. Είμαι μεταξύ αυτών οι οποίοι θεωρώ ότι εξακολουθεί αυτή η οντότητα να, είναι, να έχει αποσχιστεί από τη Σερβία και ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζουμε βεβαίως την απόσχηση από ένα ε, τέτοιο κράτος. Βέβαια, ο κύριος ε, Χισένη και ε, ο λαός του Κωσόβου ε, βιώνουν τις συνέπειες αυτής της απόσχησης γιατί ο ίδιος ο κύριος δεν εκπροσωπεί το σύνολο του λαού του Κωσόβου. Εκπροσωπεί μόνον τους αλβανόφωνους του Κωσόβου όπως γνωρίζουμε και λυπόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Επειδή ο κύριος Ισέν έκανε βέβαια λόγο για ε, ότι τα, ο πόλεμος έχει αφήσει πολλά ε, κατάλοιπα, το ίδιο ισχύει και για τους άλλους. Άρα το πρόβλημα που υπάρχει είναι να δει κανείς ε, πώς θα εξασφαλιστούν τα δικαιώματα όλων των κατοίκων του Κωσόβου, κάτι που δεν είναι διασφαλισμένο αυτή τη στιγμή και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος ε, Χισένη, ο ίδιος ίσω να μην φταίει τόσο πολύ όσο το ίδιο το σχέδιο Αχτισάρη, το απαράδεκτο σχέδιο Αχτισάρη, βάσει του οποίου γίνανε αυτά που μας είπε ο κύριος ε, Χισένη. Θα ήθελα ε, επίσης να τον ρωτήσω τι θα κάνει ο ίδιος εάν το Διεθνές Δικαστήριο βγάλει ότι είναι παράνομη η απόσχηση του Κωσόβου από την Σερβία και τελευταία, να μας εξηγήσει ποιος ο ρόλος οι Ηνωμένε Πολιτείες να έχουν μια τόσο μεγάλη στρατιωτική βάση στο Κόσοβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Eh, ευχαριστώ. Κυρία Μουνίθ, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε κύριε Χισένη που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Είπατε πολλές φορές ότι πέντε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 120 χώρες από τη διεθνή κοινότητα που ε, θεώρησαν ότι μονομερείς ανακήρυξαν εξαρτησίες χωρίς συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και χωρίς ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν συνιστούν επαρκείς βάσεις για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας και κατά τη γνώμη μου είναι σωστή αυτή η κρίση τόσων χωρών και από άποψη σταθερότητας <clears throat> γιατί η αναγνώριση του κοσυφοπεδίου χωρίς να πληρούνται οι προηγούμενες ε, προϋποθέσεις μπορεί να δημιουργήσει αστάθεια στην περιοχή. Περιμένουμε, όπως είπατε, την απόφαση, την νομική γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ερωτώ λοιπόν, με επικοδομητικό πνεύμα, τι προσδοκίες έχετε από την ε, γνωμάτευση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του ε, Δικαστηρίου θα αλλάξει τίποτα η θέση του δικαστηρίου απέναντι στις ε, χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσυφοπαίδιο εκ μέρους της χώρας σας. Ε, ποια είναι η θέση σας ως προς αυτό, τις προοπτικές μετά από τη γνωμοδότηση του δικαστηρίου. Το λόγο έχει ο κύριος Μπέλτερ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Έχω μία ερώτηση. Μια-δυο μέρες πριν έρθετε εδώ, διάβασα ένα αρκετά απεσιόδοξο άρθρο, καταθλιπτικό θα έλεγα. Πήγα μια-δυο φορές και στο κοσυφοπαίδιο και έμαθα ότι πριν από μία εβδομάδα έγινε μία σημαντική επιχείρηση της Γιούλεξ ε, για τη διερεύνηση ε, υποψίας για σκάνδαλα διαφθοράς μεγάλης κλίμακας. Διαλευκάνθηκε αυτό το σκάνδαλο γιατί από ό,τι ξέρω έγινε, έγιναν έρευνες και νομίζω είναι μπλεγμένος και ο υπουργό Υποδομών και πολύ υψηλόβαθμοι υπάλληλοι που ασχολούνται με τις εγκρίσεις για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων. Γιατί είπατε ότι σας ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή προοπτική, επιλέξατε τη δημοκρατία, οπότε η κοινή γνώμη ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει στο κοσυφοπαίδιο. Και τι γίνεται με την εικόνα της Γιούλεξ, γιατί αν η Γιούλεξ ασχολείται με την πάταξη της ε, εγκληματικότητας στο Κωσυφοπέδι, δεν ξέρω τι εντύπωση δίνει εκεί. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να εκπροσωπείτε και τις μειονότητες της χώρας σας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Μικολά για δύο λεπτά. Κύριε Υπουργέ. ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, μια σύντομη παρατήρηση. Η αναγνώριση του κράτους ε, είναι θέμα κράτους δικαίου, δεν είναι θέμα προσωπικής γνώμη. γνώμης. Αυτή είναι η ερώτησή μου και ε, είμαι βεβαίω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στο κράτος δικαίου. Έχω μία ερώτηση όσον αφορά την πολυπολιτισμική σας προσέγγιση. Επικροτώ αυτού του τύπου την ε, προσέγγιση. Είναι πολύ σημαντική για το σύνολο της περιοχής, όχι μόνο για την δική σας περιφέρεια. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με τον αποκλεισμό της ε, σερβική κοινότητας από την ε, διοικητική και ε, δικαστική διαδικασία. Έχετε μέτρο για να αυξήσετε την συμμετοχή της κοινότητας αυτής στους δύο αυτούς τομείς. Και δεύτερον, έχετε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο για να στηρίξετε την Ορθόδοξη Εκκλησία στην περιοχή. Και η τρίτη μου ερώτηση έχει να κάνει με το, με την, με το υψηλό ποσοστό ανεργίας. 40% σίγουρα δεν είναι ε, πολύ καλό. Έχετε κάποιο κοινωνικό μέτρο για να καταπολεμήσετε την ε, ανεργία. Ο κύριος Βόμποτα έχει τώρα το λόγο. Ο κύριος Βόμποτα είναι πρόεδρος της ομάδας εργασίας μας για τις σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια. Δύο λεπτά κύριε Βόμποτα. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε και αύριο στην ομάδα εργασία θα έχουμε δυνατότητα να ε, μιλήσουμε μαζί σας. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριος Βάγκελ για το θέμα των Ρώμα. Και, και στο Στρασβούργο συζητήσαμε το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό για όλες τις χώρες ε, και στη Σερβία υπάρχουν, ε, ε, υπάρχει πολύ κακή κατάσταση, αλλά για όλες τις χώρες είναι σημαντικό το θέμα της ένταξής τους. Δύο ερωτήσεις. Καταρχήν είσαστε έτοιμος, είσαστε διατεθειμένος να προωθήσετε και να βελτιώσετε τη συνεργασία ανάμεσα στις αρχές του κοσφοπεδίου και της Σερβίας σε θέματα περιβάλλοντος και άλλων, άσχετα από την αναγνώριση. Δεν μιλάω για επίπεδο κυβέρνησης, μιλάω, μιλάω για τοπικές αρχές σε τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να λυθούν όπως είναι η, απο... η αποκομιδή των απορριμμάτων κλπ. Και να επανέλθω στην ε, απόφαση του Διεθνούς ε, Δικαστηρίου, άσχετα από το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, το οποίο μάλλον ε, θα είναι ε, κάπως ασαφές όλοι θα θεωρήσουν ότι δικαιώνονται, αλλά μπορούν να ξεκινήσουν συζητήσεις με την ανεξαρτησία του κοσφοπεδίου που δεν μπορεί τώρα να ξεγίνει, ε, πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί ένα νέο πλαίσιο στην περιοχή και επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο κύριος ε, Σέβεριν. Ε, μπορεί να είναι κάπως διαφορετική η προοπτική του, αλλά πιστεύετε ότι αυτό θα πρέπει, η απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι το ξεκίνημα για νέες ε, συζητήσεις που θα βελτιώσουν την προοπτική ανεξαρτησίας, αλλά θα ε, ωφελήσουν και όλες τις ε, πλεκόμενες χώρες συμπεριλαμβανομένου του Κοσφοπεδίου και της Σερβίας. Ευχαριστούμε κύριε Σβόμποτα. Ο κύριος Κυρίλοφ για δύο λεπτά θα είναι ο τελευταίος ομιλητής στη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, όπως ε, ανέφερε ένας προλαλής ε, και εγώ διάβασα αυτό το άρθρο για τις υπόνοιες διαφθοράς κάποιων υπουργών. Είπατε ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ της Γιούλεξ ε, και των αρμόδιων αρχών. Ε, αυτή η συγκεκριμένη δράση και η δίωξη ήταν επιχείρηση της Γιούλεξ μόνο ή απόρρια συνεργασίας με τις δικές σας αρμόδιες αρχές. Επίσης, έγινε έρευνα για κάποιες ε, εγκληματικές ενέργειες και τελικά οι... κατηγορήθηκαν ε, για τρομοκρατική για τρομοκρατικές ενέργειες. Δεν ξέρω, όταν ε, συνελήθησαν αυτοί και κατηγορήθηκαν, ε, το ήξερε η Γιούλεξ ή όταν η Γιούλεξ ε, ξεκίνησε δίωξη κατά τον Υπουργό σας ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές γι' αυτό. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Κύριλοφ. Θα δώσω το λόγο στον Υπουργό, αλλά θα σας παρακαλούσα πραγματικά να τηρήσετε το δεκάλεπτο. Συνοπτικά. όσο πιο σύντομος γίνεται θα γίνω. Αλλά έχουν τεθεί τόσες ερωτήσεις που θα ήθελα λίγο περισσότερο χρόνο, αν μπορώ. Φίλε Άντριαν Σέβεριν. Έχουμε ένα όραμα, ναι. Our vision for the region is uh, cooperate closely. Ποιο είναι αυτό το όραμα. Στενή συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Αν θέλετε, ως πρελούδιο, ως προϋπόθεση για περαιτέρω ενοποίηση. Και ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να σέβεται ο ένας τον άλλον. Όχι να υπάρχει επίσημη αναγνώριση κατά ανάγκη, αλλά να σέβεται Αυτό με φέρνει και με συγχωρείτε που πηδάω από τη μία ερώτηση στην άλλη, αλλά συσχετίζονται μεταξύ τους. Με φέρνει αυτό στο θέμα της άμεσης συνέπειας της αποφάσεως του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Και των πιθανών κινήσεων στις οποίες θα προσφύγει κατά κάποιο τρόπο η Σερβία, στο σκοπεύει προφανώς. Δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα και αυτό απαντά σε κάποιες ερωτήσεις, διότι δεν είναι ακριβές ούτε σκόπιμο να προδικάσουμε το τι θα πούν τα 15 αξιότιμα μέλη του δικαστηρίου για το θέμα αυτό. Ανεξάρτητος τόσο από την έκβαση, εμείς μιλούμε για μία γνωμοδότηση που δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα έναντι ουδενός κράτους της ε, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ζήτησε τη γνωμοδότηση. Χωρίς λοιπόν να προδικάσω κάτι τέτοιο, να σας πω ότι έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο ΔΕΛΤΑ, ΔΕΛΤΑ, ΔΕΛΤΑ, διότι στο Πέδιο αποδείξαμε και παράσχαμε τα αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουμε εμπιστοσύνη στην διεθνή δικαιοσύνη και τους διεθνείς οργανισμούς απονομής δικαιοσύνης. Πολλά μπορούμε να κάνουμε σε περιφερειακό επίπεδο για να περάσουμε ένα πιο θετικό μήνυμα προς εσάς. Να διευκολύνουμε ή να απελευθερώσουμε την κίνηση, τις αγορές, το εμπόριο, Δυστυχώς όπως γνωρίζετε, η Σερβική Δημοκρατία παρεμποδίζει όλες τις εξαγωγές του κοσυφοπεδίου. Δεν εφαρμόσαμε στο μέτρο αυτό αμοιβαιότητα, για έναν απλό λόγο. Θέλαμε να αποδείξουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε στη Σερβία περισσότερο χρόνο ενώ από την άλλη πλευρά είμαστε βέβαιοι ότι κάνοντας κάτι τέτοιο, μόνο ζημία θα επιφέρουμε στις επιχειρήσεις από τις δύο πλευρές των συνόρων. If would allow exports from Kosovo. Or... Η η άλλη λύση θα μπορούσε να ήταν να, μια άλλη λύση θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ε, την εσωτερική μετακίνηση χωρίς θεωρήσεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Γιατί να χρειάζομαι βίζα για να πάω από τη μία χώρα της περιοχής στην άλλη, την Αλβανία, τη Βοσνία, το Μαυροβούνι. Πάλι με τον τρόπο αυτό θα δίναμε ένα σαφές μήνυμα ότι θέλουμε την απελευθέρωση της χορηγής θεωρήσεων με την Ένωση. Πριν το κάνουμε αυτό όμως είμαστε σε θέση να το εφαρμόσουμε σε περιφερειακό επίπεδο. Να δημιουργήσουμε ένα καθεστώς θεωρήσεων τύπου Σέγγεν στα Δυτικά Βαλκάρια. Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Αυτό που λείπει δεν είναι τα μέτρα, είναι η βούληση να εκτιμήσουμε το όραμα αυτό και να δουλέψουμε για να γίνει πραγματικότητα το όραμα. Ξέρω ότι θα αρχίσει να φωνάζει ο κύριος Αλμπερτίνη, ο καλός μου φίλος, να αρχίσω να μιλάω επί μακρόν. Για τις άλλες ερωτήσεις τώρα, εντάχει. Εκπροσωπώ όλο το λαό του Κωσυφοπεδίου. Μην κάνετε λάθος. Δεν σημαίνει ότι δεν εκπροσωπώ όλους. Όλους τους εκπροσωπώ. Όλοι οι πολίτες του Κοσμοπεδίου μετέχουν πλήρως στα θεσμικά όργανα της Δημοκρατίας του Κοσμοπεδίου. Έχουμε μέλη της σερβικής κοινότητας στο Κοινοβούλιο. Έχουμε δύο υπουργούς Σέρβους στην κυβέρνηση του Κοσμοπεδίου που αντιπροσωπεύουν όπως αρμόζει τη σερβική κοινότητα του Κωσυφοπεδίου. Η ad hoc αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, του δικού σας Κοινοβουλίου, στην, στις, ε, ε, στην έκθεσή της για τις ε, πρόσφατες εκλογές, τοπικές εκλογές, ανέφερε ότι σε ορισμένε περιοχέ, ότι σε όλες τις περιοχές είχαμε σημαντική παρουσία τη σερβική μειονότητας στις εκλογέ Από 25 με 50% σε κάποιε περιπτώσει. Δεν ξέρω αν εκπροσωπώ όλους τους πολίτε του του εκπροσωπώ ωστόσο αποτελεσματικά. Θα διαφωνήσω, εάν μου επιτρέπετε, με την κυρία Μουνής στη θέση σας ότι η ανεξαρτησία του κοσμοπεδίου δημιούργησε αστάθεια στην περιοχή. Το ανάποδο συνέβη. Ακριβώς το ανάποδο. Η ανεξαρτησία του κοσμοπεδίου επιτέλους σταθεροποίησε τα, την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Ούτε ένας Σέρβος δεν εγκατέλειψε το Κωσφοπέδιο μετά την ε, διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Το αντίθετο, πολλοί Σέρβοι επιστρέφουν στο Κοσμοπέδιο. Δεν είδαμε μείζωνα, μείζονες συγκρούσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο Κοσμοπέδιο. Αντίθετα από αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν. Άρα, το να λέμε ότι η, του, η ανεξαρτητοποίηση του κοσμοπεδίου αποσταθροποίησε την περιοχή με κάθε σεβασμό προς εσάς κυρία μου σημαίνει είτε έλλειψη ενημέρωσης έλλειψη οποιασδήποτε ενημέρωσης και ιδέας για το τι έφερε η ανεξαρτητοποίηση του κοσμοπεδίου στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων για το δικαστήριο το Διεθνές Δικαστήριο, απάντησα. Δεν θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να προδικάσω την έκβαση του δικαστηρίου. Ξέρετε ωστόσο ότι ως πολιτική. πρέπει να εξετάζουμε όλες τις πιθανότητες. Έστω ότι η απόφαση δεν είναι καθοριστική. Για μας το αποτέλεσμα της γνωμοδότησης δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι πώς θα συμπεριφερθούμε όλοι μας αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Ο φόβος και η ανησυχία μου είναι αυτό που είπα προηγουμένω. Το να έρθει η Σερβία και να επιβάλλει ε, διπλωματικά οδοφράγματα. Κάτι τέτοιο θα αυξήσει την αντιπαράθεση μεταξύ του Κωσυφοπεδίου και της Σερβίας, δεν τη μειώσει. Και ο φόβος και η ανησυχία μου είναι αυτή θα ήθελα πραγματικά να κάνω λάθος. Και αντί να πάει προς την κατεύθυνση εκείνη, το Βελιγράδι να αποφασίσει να κάτσει στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων και να μιλήσει μαζί μας. Αυτό παντά και σε μια άλλη ε, ερώτηση που τέθηκε. Βεβαίω είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε να μιλήσουμε με τη Σερβία για πολλά θέματα αμοιβαίας, ενδιαφέροντο. Ε, ε, ενδιαφέροντος και μεγάλη σημασία για την περιοχή. Γιατί οι σχέσεις μεταξύ Κοσφοπεδίου και Σερβίας σε καθημερινή βάση μετατρέπονται σταδιακά σε ένα πρόσκομα στην ευρωπαϊκή πορεία ολόκληρη της περιοχής. Τώρα, η μάχη κατά της διαφθοράς οι πρόσφατες δράσεις της Γιούλεξ και η δικαστική εξουσία του Κωσυφοπέδιο. Τι μπορώ να σας πω. Η κυβέρνηση του Κωσυφοπέδιου αγωνίζεται και επιδιώκει πάση θυσία να καταπολεμήσει την διαφθορά και το έγκλημα σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας μας. Ούτε ένας αξιωματούχος και υπάλληλος στην ε, δημόσια διοίκηση του Κοσμοπεδίου από την, τον Υπουργό μέχρι κάτω, μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο, δεν μπορεί να την γλιτώσει εάν έχει παραβεί τον νόμο. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ξεκάθαρα από αυτού, γι' αυτό έχουμε υποστηρίξει την θέσπιση ειδικών task force για την μάχη κατά της διαφθοράς. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και περισσότερες λεπτομέρειες να είχα, διότι αυτό είναι θέμα των δικαστηρίων, των ερευνητικών αρχών, δεν θα επέμβω στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και των ερευνών. Περιμένετε. Ας δούμε πρώτα ποια είναι η έκβαση Ελπίζω να μπορέσουμε να χτυπήσουμε όσο καλύτερα γίνεται τη διαφθορά και το έγκλημα που βρίσκεται δυστυχώς σε όλη την περιοχή. Μην, δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε, να χτυπήσουμε το οργανωμένο έγκλημα μόνο στο Κωσυφοπέδιο, αν δεν το χτυπήσουμε και στη Σερβία, την Αλβανία, το Μαυροβούνι, τη Βοσνία κτλ. συν, συνεργάζονται πολύ καλά, ξέρετε, οι οργανωμένοι εγκληματίε μεταξύ τους. Πρέπει να συνεργαστούμε ω αρχές στην Πριστίνα και στο Βελιγράδι για να χτυπήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Δεν μπορείτε να πείτε ότι θα χτυπήσετε το έγκλημα όταν αποκλείσουμε, αν αποκλείουμε από τις προσπάθειες αυτές το κοσμοπέδιο. Και η Σερβία κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει τη συμμετοχή του κοσμοπεδίου εκεί. Υπήρχε και μια άλλη ερώτηση που βασικά αφορούσε την πολυπολιτισμική διάσταση του κοσμοπεδίου και τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει την ε, πολυ... Ε, πολυπιτισμικότητα. Μην το αμφιβάλλετε, το θέλουμε αυτό πραγματικά. Πρέπει να διαφωνήσω με τη δήλωσή σας χρησιμοποιήσετε τον όρο αποκλεισμό τη σερβική κοινότητα. Ποτέ δεν το κάναμε αυτό. Ποτέ δεν αποκλείσαμε τη σερβική κοινότητα από τι κοινέ μα προσπάθειε. Καλέσαμε επανειλημμένα τη σερβική κοινότητα να συνεργαστεί μαζί μας στις προσπάθειες να επιβάλλουμε μια πολυπολιτισμική διάσταση του κοσυφοπεδίου. Όλο και περισσότεροι Σέρβοι έρχονται προς εμάς. Αυτό είναι καλά νέα. Για να μην σας πω ότι όλοι θα έρθουν τελικά. Διότι αναγνώρισαν ότι και το λέω αυτό με, δυστυχώς με μεγάλη επιφύλαξη. Αναγνώρισαν ότι το Βελιγράδι μόνο κουβεντιάζει, μιλάει, δεν κάνει τίποτα για να βελτιώσει τις συνθήκες των, ε, της ερευνικής κοινότητας του Κοσμοπέδιο. Το Βελιγράδι χρησιμοποιεί τη ερευνική κοινότητα του Κοσμοπέδιο ως άλοθη για να αποσταθεροποιήσει βαθιά το κοσμοπέδιο, ούτως ώστε εν τέλει να έχει ένα πρόσχημα για να επαναφέρει τις διαπραγματεύσεις, διαπραγματεύσεις για το καθεστώς του κοσμοπεδίου. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Είναι ανεξάρτητο το Κόσοβο. Αυτό είναι μια διαδικασία χωρίς επιστροφή. Κλείνω με μια θετική νότα. Ελπίζω μετά το δουδουδού το Βελιγράδι να μετάσχει στις κοινέ προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε ένα κλίμα αμοιβέ κατανόησης και να συνεργαστεί μαζί μας για την ειρήνη και την, ε, και την ευρωπαϊκή προεπτική όλης της περιοχής. Σας ευχαριστώ. Συμφω... Δεχόμαστε και συμμεριζόμαστε την ευχή σε αυτή, κύριε Υπουργέ. Θα τα πούμε σε μια επόμενη συνάντησή μας, όπου ελπίζω και εγώ και όλοι μας, όχι μόνο εσείς, να έχουμε εικόνα για τις εξερίξεις προς το κράτος δικαίου, την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα σας και την προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστούμε εκ νέου, σα αποχαιρετούμε και ελπίζω να το πούμε σύντομα. Κύριε Danjean, ελάτε στη... στο βήμα για να προεδρεύσετε στην ανταλλαγή απόψεων για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της ΚΕΠΑ στην περίοδο μετά την Δυτικό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά κρατάμε δύο-τρία λεπτά για να μπορέσουν οι συνάδελφοι που έχουν άλλες δουλειές να φύγουν ma il tempo è così tiranno che ci obbliga a proseguire la Έχουμε όμως υποχρέωση να προχωρήσουμε. Εισαγωγικά, στις 31 Μαΐου του 2000, ε, Μαρτίου συγγνώμη, του 2010, η Προεδρία του Συμβουλίου της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης ΔΕΕ δήλωσε την πρόθεσή της την πρόταση των 10 κρατών μελών να καταγγείλουν την ε, συμφωνία, τη συνθήκη ΔΕ και να θέσουν, να, να οδηγήσουν στη λήξη μέσα στον Ιούνιο της ΔΕ και της συνέλευσής Η δήλωση αυτή ακολουθήθηκε από μια κοινοβουλευτική συζήτηση στην Γαλλική Κερουσία και στη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλου για τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων που είναι προσαρτημένο στη συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να βρουν συμφωνία για να εξασφαλίσουν και αποτελεσματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο στην, πολιτική ασφάλεια, στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Το θέμα αυτό ήδη εξετάστηκε και τέθηκε και κλεισμένων των θυρών στη συνάντηση της 27ης Απριλίου του 10 και από την ομάδα παρακολούθησης για τα Εθνικά Κοινοβούλια που όπως ε, ξέρετε στην Επιτροπή Ασφάλειας και από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Ο κύριος Νταφ ήταν παρόν και στις δύο συναντήσεις, στην Υποεπιτροπή Ασφάλειας και στην Επιτροπή Παρακολούθησης και μπορεί να μας παρουσιάσει και μια σειρά μοντέλων ε, κοινοβουλευτικής παρακολούθησης θεμάτων ασφάλειας και άμυνας Εμεί πρέπει ω Κοινοβούλιο να επιλέξουμε ποια οδό θέλουμε μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό εισαγωγικά. Θα δώσω τώρα το λόγο στο συνάδελφο κύριο Ντανζάν, πρόεδρο τη Υποεπιτροπή Ασφάλεια και Αμύνα και κατόπιν στον κύριο Νταφ για να μας παρουσιάσουν τα επιχειρήματα που περιέγραψα. Κύριε Ντανζάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι λακωνικότατος γιατί τα είπατε όλα και κάνατε μία πολύ σωστή ανακεφαλαίωση της κατάστασης. Θα πρέπει πολύ σύντομα να διερευνήσουμε τα διάφορα σενάρια στις συζητήσεις που θα έχουμε με τους εθνικούς βουλευτές και σε δέκα περίπου μέρες θα έχουμε μια συνεδρίαση πρόεδρη των Εθνικών Κοινοβουλίο μαζί με τον πρόεδρο Μπούζεκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέχρι τότε ελπίζω να έχουν κάποιες ενδείξεις για τους προσανατολισμούς μας ώστε να είναι πλούσιες οι συζητήσεις αυτές. Οι συνάδελφοί μας από τις Εθνικές Βουλές νομίζω ότι θα εγκύψει το θέμα αυτό πολύ γρήγορα και όπως είπατε ήδη η Γαλλική Γερουσία και η Βρετανική Βουλή των Αντιπροσώπων ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό και έλαβαν θέση. Και μάλιστα θα γίνει και μια ειδική, ειδικευμένη κοζάκ με τη συμμετοχή έξι ε, εθνικών βουλευτών και έξι, ευρωβουλευ... έξι εθνικών βουλευτών από κάθε κοινοβούλιο και έξι ευρωβουλευτών για ε, συνεδρίαση δύο φορές το χρόνο. Βέβαια, θα είναι λίγοι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολλοί των Εθνικών Κοινοβουλίων. Παρόλο που τον άρθρο 36 της ε, συνθήκης μας δίνει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ε, συνέχεια το κοινοβουλευτικό έλεγχο της ΚΕΠΑ αλλά φαίνεται ότι θα καταιγιστεί το Κοινοβούλιο από εθνικούς βουλευτές για το θέμα αυτό. Εγώ είμαι υπέρ μιας ρεαλιστικής και λειτουργικής λύσης. Α μην ξεχνούμε ότι ένα από του λόγου που δικαιολογούν τη διάλυση τη ΔΕΕ και της κοινοβουλευτική συνέλευση είναι το θέμα του κόστου και της λειτουργικότητα. Θα πρέπει και αυτό λοιπόν να το λάβουμε υπόψη στι διάφορε προτάσει που θα αναλύσουμε. Σε αδρες γραμμε γραμμές έχουμε τρει-τέσσερι εναλλακτικέ λύσει που θα πρέπει να διερευνήσουμε, αλλά θα δώσω το λόγο στον Άντριου Νταφ για να μα τι παρουσιάσει, γιατί έκανε μια πολύ σημαντική προεργασία σύνθεσης αυτών των τεσσάρων εναλλακτικών λύσεων. Κύριε Ντάφ, ε, περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία την παρουσίασή σας. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί μου δίνετε ευκαιρία να συνεχίσουμε μια συζήτηση που άρχισε πριν από λίγο για τη βελτίωση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Και μάλιστα η ίδια συνθήκη μας υποχρεώνει να βελτιώσουμε την συνεργασία μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δεν είναι θέμα διακριτικής μας ευχέρειας. Είναι υποχρέωσή μας. Και είναι πολύ σωστή αυτή η συμπερίληψη της ε, σχετικής ρήτρα στη συνθήκη. Γιατί ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητές μας σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων ή θέματα πολιτικής εσωτερικής ασφάλειας, αλλά και κοινή ε, εξωτερικής πολιτικής ε, και πολιτικής ε, ασφάλειας και άμυνας. Η ΚΕΠΑ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος τομέας και για τα εθνικά κοινοβούλια και για αιώνες ολόκληρους ε, την ε, κρατούσαν ως φυλαχτό. Και μάλιστα στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε ε, ιδιαίτερες δυνατότητες ε, να καταθέσει την εμπειρογνωμοσύνη του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ε, και ασφάλειας. Στο μεταξύ όμως και εμείς γίναμε πιο ειδικοί για τα θέματα αυτά και σε κάποιο βαθμό εκφράστηκε κάποια ζήλια από τα Εθνικά Κοινοβούλια εξαιτία τη αυξανόμενη σημασία που λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα θέματα αυτά. Μάλιστα, η ίδια συνθήκη προβλέπει ότι θα πρέπει να καθορίσουμε τον, τη μορφή τη διακοινοβουλευτική συνεργασία. Αποκινούμε τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δηλαδή, τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν για το τι δρόμο θα ακολουθήσουν. Μάλιστα, η, με αποσταθεροποίησε κάπως ε, η, η απόφαση το, και της Γαλλικής Γερουσίας και της ε, Βρετανικής Βουλής των Αντιπροσώπων να συνεχίσουν μόνο, από μόνος τους χωρίς, αν δεν υπάρχει κανονική διαβούλευση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Στα φόρα που έχουμε, έχουμε τους προέδρους των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων με τον πρόεδρο Μπούζεκ. Έχουμε την ΚΟΖΑΚ και έχουμε και την ΚΟΦΑΚ που είναι η συνδιάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σε ό,τι αφορά το έγγραφο που συνέταξα για την ομάδα εργασίας. Εγώ εντόπισα τρεις ε, εναλλακτικές λύσεις. Η πρώτη είναι μια ελαστική μορφή της διακοινοβουλευτικής συνάντησης που είχαμε στο παρελθόν, που θα γίνεται υπό τη δική μας οργάνωση και καθοδήγηση. Εμείς θα καθορίζουμε την ημερήσια διάταξη και θα προσκαλούμε τους εκπροσώπους των Αθηνικών Κοινοβουλίων, αν το επιθυμούν να έλθουν, γιατί υπήρξαν πολλά παράπονα βέβαια από, από τα Εθνικά Κοινοβούλια για αυτή τη μορφή συνεργασία. Ε, παραπονέθηκαν για την κακή διοργάνωση, η δομή. Τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν παρακολουθούν ιδιαίτερα αυτές τις συνεδριάσεις. Αυτή είναι η πρώτη μορφή ελαστική συνεργασία, Η δεύτερη εναλλακτική λύση είναι αυτή που προτιμούν η Γαλλική Γερουσία και η παλιά βουλή των αντιπροσώπων. Είναι η ίδρυση μια νέα ειδικευμένη ΚΟΖΑΚ. Μια ΚΟΖΑΚ που θα είναι αφιερωμένη σε θέματα και πά. Ο πρόεδρος Ντονζόν ήδη μας ε, παρέθεσε κάποια μειονεκτήματα μιας τέτοια νέα οργάνωση και από άποψη κόστου και από άποψη της ε, πολύ μικρή συμμετοχή εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εγώ πιστεύω ότι μια τέτοια κοζάκα ε, δεν αντικατοπτρίζει πιστά το πνεύμα της συνθήκης. Η συνθήκη έχει σταθεροποιήσει τις προεδρίες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για θέματα και πάει γιατί έχουμε πλέον ένα μόνιμο πρόσωπο, πρόεδρο και καθορίστηκε και ο ρόλος της Καθρινάστον που θα είναι η μόνιμη εκπρόσωπος του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών. Και μάλιστα και η, Τρόικα, η λειτουργία της Τρόικας έχει σχεδόν ε, εξαφανιστεί. σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Και νομίζω ότι και από κοινοβουλευτική άποψη θα πρέπει να υπάρχει αντανάκλαση της νέας κατάστασης με τη μόνιμη Προεδρία. Σε ό,τι αφορά το εκτελεστικό τμήμα του θεσμικού πλαισίου. Η τρίτη εναλλακτική είναι αυτή που προτιμώ εγώ και είναι η πρόταση για μικτές συνεδριάσεις των Επιτροπών με από κοινού διοργάνωση δική μας και της α, εκπεριτροπής Προεδρίας. Του Κοινοβουλίου δηλαδή της εκπεριτροπής Προεδρίας, της χώρας που ασκεί κάθε εξάμενο την Προεδρία. Μία τέτοια εναλλακτική λύση δεν απαιτεί την ίδρυση μιας νέας γραμματείας και είναι η φθηνότερη λύση, γιατί όλα θα γίνονται στις Βρυξέλλες, ε, τις δαπάνες θα τις καταβάλει το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ίσως χρειαστούμε δύο τέτοιες συναντήσεις το χρόνο, μία κάθε εξάμεινο. Νομίζω ότι αρκούν. Στην πρώτη θα επικεντρωνόμαστε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και στη δεύτερη σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Οι μικτές αυτές συνεδριάσεις θα εξετάζουν και εκθέσεις συζητών για τα πιο επίκαιρα θέματα, τα πιο αφλέγοντα, καθώς και τις απόψεις μας για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ΚΕΠΑ και για την επιτυχία ή αποτυχία των επιχειρήσεων της ΚΕΠΑ. Επίσης, τέτοιες μεκτές συνεδριάσεις θα περιμένουν από την Κάθρια Άστον και τον πρόεδρο Βαρερόν τακτικές εμφανίσεις ε, στις ε, συνεδριάσεις αυτές τις μικτές, προκειμένου να δίνουν απαντήσεις ε, σε απορίες και ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών και των Εθνικών Βουλευτών. Μάλιστα τέτοιου είδους συναντήσεις θα έχουν σημαντική απήχηση και θα προβάλλονται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα μας βοηθήσουν στο να γεφυρώσουμε κάπως ε, το δημοκρατικό χάσμα ή το δημοκρατικό έλλειμμα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και της μόνιμης Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στην οργάνωση αυτή θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και εκπροσώπους των κοινοβουλίων τρίτων χωρών και μάλιστα θα μπορούσαμε να προσκαλέσουμε ίσως και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που από ό,τι ξέρω και αυτός αναζητά το κατάλληλο φόρουμ εντός α, ε, της δομής αυτής για να έχει ένα βήμα να μιλήσει. Βέβαια θα πρέπει να αποσαφιλιστούν οι σχέσεις αυτής της Μικτής Επιτροπής με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ. Φυσικά θα συμμετέχουν ε, ευρωβουλευτές από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικοί βουλευτέ, αλλά δεν θα είναι ένα σώμα που θα καταρτίζει ψηφίσματα. Αυτές οι τη Μικτής Επιτροπής δεν ε, θα εγκύπτουν κατά ανάγκη σε συγκεκριμένα κείμενα, ούτε θα χρειάζεται να, να λαμβάνονται αποφάσεις. Νομίζω ότι αυτή η τρίτη εναλλακτική λύση είναι και πιο ελκυστική για μας, αλλά και για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Όπως είπε ο κύριος Δανζόν, καλό θα είναι να σπεύσουμε και να λάβουμε μία απόφαση για το θέμα αυτό, αλλιώς θα δημιουργηθεί ένα κενό δικαίου που θα γεφυρωθεί από μια αυθόρμητη δράση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε εδώ και το μνημόνιο συνεννόησης που προσπαθούμε να συνυπογράψουμε με την Κάθριν Άστον. Σε ό,τι αφορά τη δέσμευσή της να δίνει το παρόν τακτικά σε τέτοιου είδους ε, κοινέ συνεδριάσεις, μικτές συνεδριάσεις και να έχουμε επίσης τακτικές επαφές ε, με τον πρόεδρο Βαν Ευχαριστώ. Μπάστα. Ευχαριστούμε. Ο κ. Γκάλερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη πριν τη θέση σε ισχύ της συνθήκη της Λισαβόνας πάντα έλεγε ότι είμαστε το μόνο κοινοβουλευτικό όργανο, το μόνο ε, υπερεθνικό που μπορεί να εποπτεύει την εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας και με την ε, θέση σε ισχύ της συνθήκης της αυτό είναι πιο σαφές. Η... Έγινε η απόφαση να αντικατασταθεί η Ένωση της Δυτικής Ευρώπης και αυτό νομίζω ότι είναι σαφές μήνυμα. Ιδέα. αλλά αυτό ήδη το είπαμε στην έκθεση Donjon. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να συμπεριλάβουμε στη δουλειά μας ε, την πυρογνωμοσύνη και τη δουλειά των ε, εθνικών βουλευτών. Πιστεύω ότι στο δικό μας πλαίσιο υπάρχει καλύτερη δυνατότητα να προωθήσουμε περαιτέρω την, ε, ε, πολιτική, την πολιτική άμυνας και ασφαλείας της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Και πιστεύω ότι καλό θα είναι να υποβάλουμε συγκεκριμένε προτάσεις. Δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά να πω ότι επί της αρχής συμφωνώ με αυτό που πρότεινε ο συνάδελφος Ντάφ. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πολύ καλή πρόταση στους ε, συναδέλφους στα Εθνικά Κοινοβούλια και από κοινού. Να ε, εφαρμόσουμε ό,τι καλύτερο για την ε, πολιτική ασφαλείας και άμυνας της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σεβερίν. Δύο λεπτά. Πρόεδρε, εδώ και εβδομάδες προσπαθώ να συναντήσω τον κύριο Ντανζάν και τον κύριο Νταφ για να προσπαθήσουμε να έχουμε μια δια ο, διομαδική προσέγγιση στο θέμα αυτό που αφορά και την οπτική γωνία της συνεργασίας με τα Εθνικά Κοινοβούλια και την προσπάθεια να υπάρξει δημοκρατική νομιμοποίηση σε ένα σημαντικό στόχο που έχουμε. Την πρόθεση κοινών πολιτικών ασφάλειας και άμυνας για να είμαι σύντομος. Δεν πιστεύω ότι σε δύο λεπτά μπορούμε να λύσουμε το θέμα. Η λύση που προτείνει ο κύριος, η, τρί, η, η τρίτη λύση του κυρίου Νταφ είναι η πιο ελκυστική με δύο σχόλια. Ένα, να αν φέρουμε όλα τα μέλη των, Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων, θα πρέπει να συναντηθούμε σε ποδοσφαιρικό στάδιο. Επίσης, δεν πρέπει να λάβουμε υπόψη την διάλυση, το γεγονό ότι στην Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν μέλη που δεν είναι μέλη της, Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν καλύπτονται από τη δική μας το δικό μας κανονισμό. Εγώ θα πρότεινα λοιπόν να συναντηθεί μια μικρή ομάδα συναδέλφων για να από πολλές ομάδες κατά προτίμηση ώστε μαζί με κάποιους εκπροσώπους της υποεξαφάνιση κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τρίτη εναλλακτική πρόταση του κυρίου Νταφ για να ή κάτι παρόμοιο που θα επιτρέψει και σε χώρες που είναι σημαντικές για την ασφάλεια και την άμυνά μας και δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετάσχουν. Ευχαριστώ κύριε Σεβερίν. Η... η κυρία Λέζινγκ, δύο λεπτά. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο Ντάφε για τις ε, προτάσεις του. Δεν είναι πολύ εύκολο να βρούμε ε, χρήσιμες και εφαρμόσιμες λύσεις. Συμφωνούμε ότι στηρίζουμε τη λύση Γ, ωστόσο θα θέλαμε κάποιες διευκρινήσεις. η πολιτική μας ομάδα θέλει όχι μόνο να συμμετέχουν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα του κάθε κοινοβουλίου, αλλά και οι μικρότερες πολιτικές ομάδες. Διότι μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει διαφανής και δημοκρατικός έλεγχος ε, της ΚΕΠΑ. Και η συναντήσεις δύο φορές το χρόνο βρίσκουμε ότι είναι πολύ λίγες. Ε, από την ε, εμπειρία μου γνωρίζω πόσο διαφορετικά είναι τα θέματα που μπορούν να συζητηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ε, είναι απαραίτητο να συζητιόνται αυτά για να είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κρίσεων. Δεν αρκούν λοιπόν δύο συναντήσεις το χρόνο. Προτείνουμε μηνιές συναντήσεις ή διμηνιές. Γνωρίζουμε ότι η διαθεσιμότητα της ε, είπα της εκπροσώπου ή του κυρίου ε, Φανρόμπη δεν μπορεί ε, να διασφαλίζεται κάθε φορά. Ευχαριστώ κύριε Γιαννάκου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Άντριου Νταφ για την συνοπτική του παρουσίαση και νομίζω ότι από την έκθεση του, τη μικρή του έκθεση είναι αβίαστο το συμπέρασμα. Η λύση τρία, κύριε Πρόεδρε, είναι η σωστότερη όλων. Ε, καταρχήν, ε, οι συνεδριάσεις πρέπει να γίνονται στις Βρυξέλλες. Εμείς διαθέτουμε το σύστημα και νομίζω ότι σε αυτές τις συνεδριάσεις μπορούμε να καλέσουμε τρία μέλη από το κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο και λέω τρία γιατί περίπου οι πολιτικές δυνάμεις χρειάζονται τρία μέλη για να είναι όλες εκπροσωπούμενες ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε εδώ τις συνεδριάσεις με τη συμμετοχή του συνόλου των μελών ε, της ε, Επιτροπής Εξωτερικών. Νομίζω ότι δύο συνεδριάσεις το χρόνο και κάποια preparatory meetings, εάν ορίζουμε εισηγητές, επαρκούν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έτσι κι αλλιώς τα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, κύριε Πρόεδρε, τα κρατούν οι κυβερνήσεις με τον πιο σκληρό τρόπο στα χέρια τους και συνήθως ενημερώνουν τα κοινοβούλια. Εμείς θα μπορούσαμε βέβαια μέσω διαδικασιών, εισηγητών κλπ. να δώσουμε διάφορες κατευθύνσεις. Τώρα για τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση Κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω εκλεγεί τέσσερι φορέ στο Εθνικό Κοινοβούλιο και ήμουν μέλο και στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο τη Ευρώπη και παντού. Δεν έχει νόημα η συντήρηση τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Κανένα νόημα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, ανάλογα με τα θέματα, να καλούμε και αντιστοίχου βουλευτέ από τι αντίστοιχε επιτροπέ χωρών που δεν είναι μέλη, αλλά που συζητούμε διάφορα θέματα δικά τους και άλλωστε είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής εποχής. Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών. Νομίζω λοιπόν ότι ούτε η ΚΟΖΑΚ ούτε κάτι διαφορετικό καινούριο θα έχει κόστος και δεν θα εξυπηρετήσει. Ο καλύτερος τρόπος είναι η λύση 3 όπως την πρότεινε ο κύριος Νταφ. Ευχαριστώ κύριε Γιαννάκο. κύριος Πάσκο και αντιπρόεδρος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω το θέμα αυτό πρέπει να το δούμε με σαφή, με κάποιες σαφείς θέσεις, ξεκινώντας από την πραγματικότητα. Ένα, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μία ένταση μεταξύ του ότι εμείς ανήκουμε σε ένα κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, ενώ οι αποφάσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας συνεχίζουν να είναι εθνικές αρμοδιότητες. Τα εθνικά κοινοβούλια πιστεύω ότι αυτά είναι που θα έχουν τον τελικό λόγο. Αλλά θα έχουν τον τελικό λόγο για την εθνική συνεισφορά σε ένα που ολοένα και περισσότερο γίνεται σε, μια, ένα τομέα που ολοένα και περισσότερο γίνεται πολυεθνική ε, δραστηριότητα. Μπορεί να μην είναι και όταν δεν είναι, ε, μπορεί να μην είναι πολιτική, να μην είναι αποκλειστικά ε, στρατιωτική να είναι πολιτικο-στρατιωτική και ότι δεν μπορείς να έχεις σε μια τέτοια προσέγγιση μια εσωστρεφή ε, στάση. Η βάση της προσέγγισης μας νομίζω αυτή πρέπει να είναι. Και οι προτάσεις που παρουσίασε ο κύριος Νταφ ε, είναι πολύ σοφές. Να προσθέσω μόνο κάτι είναι αναγκαίο να λάβουμε υπόψη την ανάγκη για μια ad hoc ταχεία διαβούλευση. Διότι συχνά αυτό δημιουργεί προβλήματα, όχι οι τακτικές ε, συναντήσεις που γίνονται και ξαναγίνονται και ξαναγίνονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πάσκου. Κυρία Νικολά έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να τηρήσουμε όχι μόνο το γράμμα, αλλά και το πνεύμα της συνθήκης. Θα ήθελα να επανέλθω εδώ στο άρθρο 9 που προβλέπει με σαφήνεια ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να οργανωθεί σε διαβούλευση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι μια απόφαση που θα τη λάβουμε μερικώς εμείς, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε προηγουμένω διαβουλεύσει με τα εθνικά κοινοβούλια που θα συμβάλλουν και είναι αρμόδια για το δεύτερο μέρο τη απόφαση. Από κοινού θα ληφθεί αυτή η απόφαση. Επίση, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην συνεργασία σε στρατιωτικά και μη στρατιωτικά θέματα. Ίσως χρειαζόμαστε ένα πληρέστερο έγγραφο, ξεκινώντας από το έγγραφο εργασίας του Άντριου Νταφ, αλλά εμπλουτίζοντάς το με μία σε αυτές τις ad hoc διαβουλεύσεις. Και μου ήταν το συντομότερο δυνατό να διοργανώσουμε μία συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια, γιατί το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Και υπάρχει ευαισθησία εκ μέρους των Εθνικών Κοινοβουλίων, ίσως υπάρχουν και διαφορετικές ερμηνείες της συνθήκης και γι' αυτό πολλοί βουλευτές εθνικοί θεωρούν ότι έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για αυτό το τομέα. Γι' αυτό και με υπέρ μια στενή συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ήρθε η ώρα να εγκαταλείψουμε πια την ε, κοινοβουλευτική συνέλευση της ΔΕ και να λάβουμε αποφάσεις για μετά το 2011. Σας ευχαριστώ. Το λόγο για δύο λεπτά ο κύριος Γουαλτιέρη. Ευχαριστώ. Και εγώ εκτιμώ ιδιαίτερος ε, το έγγραφο του κυρίου Νταφ που διευκρινίζει ένα κέριο θέμα σε θεσμικό επίπεδο. Γιατί έχουμε αφενός την θεσμική, την διαδικασία λήψη απόφασης για την ΚΕΠΑ και άλλο θέμα είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Άλλο η απόφαση και άλλο ο κοινοβουλευτικός έλεγχος με βάση το άρθρο 36 αρμόδιο για το κοινοβουλευτικό έλεγχο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και υπάρχει και ο δημοσιονομικός έλεγχος ε, των ε, μη στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΕΠΑ. Και για αυτούς τους λόγους, αλλά και για λόγους οικονομίας, θεωρώ ότι είναι ανέφικτη λύση που προτείνει η Γαλλική Γερουσία. Και συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι θα πρέπει περαιτέρω να αναπτύξουμε την τρίτη εναλλακτική λύση. Αυτή να προωθήσουμε, αλλά ταυτόχρονα, όπως είπε ο κύριος Σεβερίν, να διαφυλάξουμε τη σημαντική πτυχή της ΔΕ που προϋποθέτει συμμετοχή και τρίτων χωρών. Επίσης, δεν αναφέρεται συγκεκριμένα ότι το άρθρο 10 του πρώτου πρωτοκόλου ε, αναφέρεται στη δεύτερη εναλλακτική λύση. Ότι δηλαδή η δεύτερη εναλλακτική λύση, η λύση Β είναι αυτή της, της πλανόδιας Κοζάκ, αλλά χάρη και στην τρίτη εναλλακτική λύση θα μπορούσαμε να περιλάβουμε κάποια στοιχεία που θα συνδυάζουν το μοντέλο που προτείνει ο κύριος Νταφ με την πρόταση για την ειδικευμένη Κοζάκ. Εκεί υπάρχει ένα περιθώριο ελιγμό και επεξεργασίας χωρίς όμως να υποσκάπτουμε τη βασική απέτηση που είναι η συνεργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό που θα γίνεται στις Βρυξέλλες με βάση μια γραμματεία που θα εδρεύει εδώ. και όχι μιας πλανόδιας κοζάκ. Οπότε, η εναλλακτική λύση 3 κατά τη γνώμη μου είναι η πιο δόκιμη. Θα μπορούσαμε να βαθύνουμε σε αυτή και να δούμε τι αντιρρήσεις ή τι ενστάσεις έχουν τα Εθνικά Κοινοβούλια ως προς αυτό. Σας ευχαριστούμε κύριε Γουαλτιέρη. Ο τελευταίος ομιλητής στη συζήτηση θα είναι ο συμπρόεδρος αυτής της ε, συνεδρίασης, αλλά πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, ο κύριος Νταμζόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα σχόλιά σας. Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση υπέρ της τρίτης εναλλακτικής λύσης από το έγγραφο του κυρίου Νταφ. Αυτή είναι η λύση που θέλουμε να εκλεπτύνουμε, να διευκρινίσουμε, να αναπτύξουμε σε ό,τι αφορά τον τρόπο συμμετοχής. Υπάρχει φυσικά και το φλέγο ζήτημα για τους συναδέλφους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της ΔΕΕ, το θέμα της συμμετοχής των τρίτων χωρών. Επίσης θα ήθελα να επισήσω την προσοχή σας ότι 24 τρίτες χώρες αυτή τη στιγμή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις στην ΚΕΠΑ. Περισσότερες δηλαδή από αυτές που συμμετέχουν στη ΔΕΕ. Οπότε όλες αυτές θα νομιμοποιούνται κάποια στιγμή. Ανάλογα και με τη συχνότητα των συνεδριάσεων. Και νομίζω ότι μία συνεδρία στο εξάμεινο είναι λογικός ρυθμός. Γιατί υπάρχει δυσκολία και επιμελητίας αλλά και πολιτική δυσκολία για να συγκαλέσουμε Μία τέτοια συνεδρίαση με τόσο σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα. Νομίζω δύο συνεδριάσεις το χρόνο είναι αρκετές. Και σε περίπτωση κρίση, έκτακτης περίπτωση. μπορούμε ίσως ε, να έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση σε πιο περιορισμένη σύνθεση. Αλλά νομίζω ότι μία φορά το εξάμεινο μπορούμε να συζητούμε θέματα επιχειρήσεων και πά. Αλλά σε κάθε επιχείρηση έχουμε και καμιά δεκαριά τρίτες χώρες που συμμετέχουν σε τέτοιες επιχειρήσεις. Οπότε θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Συμφωνώ με τους κυρίους Πάσκου και Σεβερίν. Αυτό που με εντυπωσίασε στη συζήτηση στη Γαλλική Γερουσία ήταν η άγνοια πολλών εθνικών βουλευτών για τη φύση της ΚΕΠΑ και των επιχειρήσεων ΚΕΠΑ. Γιατί περισσότερο εστιάστηκα σε στρατιωτικά θέματα που είναι εθνική αρμοδιότητα και για τα θέματα του προσωπικού αλλά και για τα θέματα του δημοσιονομικά. Από τις 13 όμως επιχειρήσεις και ΠΑ, 10 είναι μη στρατιωτικές, τρεις μόνο είναι στρατιωτικές. Και, και για τη Γεωργία και για το πρώτο πιο σημαντικές ε, ήταν μη στρατιωτικές. Θα πρέπει λοιπόν να ενημερώσουμε τους ε, συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια για τις δυνατότητες αυτές. Και φυσικά θέλουμε να συμμετέχουμε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο αυτών των επιχειρήσεων που είναι πολύ περισσότερο μη στρατιωτικές παρά στρατιωτικές. Θα πρέπει όμως να συμπληρώσουμε αυτή την έλλειψη γνώσεων και την άγνοια που χαρακτηρίζει μερικές φορές τους βουλευτές ως προς το χαρακτήρα αυτών των επιχειρήσεων. Καλό θα ήταν και οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να ορίσουν αρμόδιους ε, για το θέμα αυτό, ώστε να μπορούμε να συναντιόμαστε γρήγορα και να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες ενδείξεις και προσανατολισμούς προς τον πρόεδρο Μπούζα και να τις μεταφέρει στους ομολόγους του από τα Εθνικά Κοινοβούλια και ταυτόχρονα να δούμε πώς θα δρομολογηθούν οι συζητήσεις και με τους ομολόγους από τις κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Ο κύριος Νταφ Συμφωνώ απολύτως. Κύριε Ντονζόν, να συμφωνήσω ότι η Διευθύνουσα Ομάδα για τις για τα Εθνικά Κοινοβούλια θα συναντηθεί ε, Τετάρτη πρωί, ο πρόεδρος θα είναι, πέμπτη πρωί, συγγνώμη, ο πρόεδρος Μπουζεκ θα είναι εκεί, θα συζητηθεί το θέμα αυτό, θα τους αναφέρω το αποτέλεσμα της συζήτησης αυτής και θα προωθήσουμε γρήγορα το θέμα. Ε, όσον αφορά την, την επιχειρησιακή πλευρά στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Με πολύ καλό και συνθετικό τρόπο παρουσιάστηκε η έκβαση της συνάντησης αυτής. Σας ευχαριστώ για την, το συγκεκριμένο τρόπο και την ικανότητα σύνθεσης που εκδηλώσατε και, και αναφέρατε. Πιστεύω ότι μπορούμε να κλείσουμε το κομμάτι αυτή, αυτό της συνάντησης. με την υποχρέωση από πλευρά μου να συνοψίσω τη συζήτηση σε μία επιστολή που θα αποστείλω από κοινού προς τον πρόεδρο κύριο Μπούζεκ για να έχει επίγνωση της συζήτησης πριν τη συνάντηση που θα γίνει 15 Μαΐου με τους πρόεδρους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό θα είναι ένα από τα υποσυζήτηση ζητήματα. Επιστολή όπου θα περιλαμβάνουμε την κυρίαρχη ε, άποψη μεταξύ ημών, την επιλογή της τρίτης εναλλακτικής λύσης που, μεταξύ αυτών που πρότεινε ο κύριος Νταβ. Ε, στην λύση αυτή νομίζω στράφηκαν οι περισσότερες ε, θέσεις των συναδέλφων, αν και όλοι τόνισαν την ανάγκη να την χτενίσουν κάπως και να την κάνουν κάπου περισσότερο συμβατή σε ένα πλαίσιο πιο σύνθετο από αυτό που είχαμε αρχικά υπόψη μας. Προτείνω λοιπόν το είπατε και εσείς, συμφωνώ και εγώ, ότι πρέπει να υπάρξει μια ομάδα εργασία μαζί με την ΣΕΝΤΕ, την Υποεπιτροπή, για την ανάλυση του θέματος και με έναν διάλογο ενδεχόμενα με τις αντίστοιχες επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, είτε εξωτερικών υποθέσεων είτε ασφάλειας και άμυνας. Ωραία. Να προχωρήσουμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη. Έχουμε την ανταλλαγή απόψεων